Vayan ocupando Καθίστε παρακαλώ και να ετοιμάσετε και τις καρτούλες. Έχω την ευχαρίστηση να σας πληροφορήσω ότι ε, είναι παρούσα εδώ μια επίσημη αντιπροσωπεία που αποτελείται από θρησκευτικού ηγέτες χριστιανούς ιδιαιτέρως της Μέσης Ανατολής από το Ιράκ και από τον Λίβανο είναι μεταξύ μας εδώ γνωρίζουμε καλά πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση για τους χριστιανούς στην περιοχή αυτή και θα θέλαμε να τους εκφράσουμε την υποστήριξή μας, την πλήρη μας υποστήριξη. Σας καλωσορίζουμε πάντως εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.